και να βάλουμε ποια θέματα έχουν προτεραιότητα για μας μέσω υποχρεωτικών απαιτήσεων και να μην βασιζόμαστε επί ρητρών που χρησιμοποιούνται θελοντικά. Μερσή κύριε Τέιλορ. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές ο κύριος Βαντάλεν για 1,5 λεπτό.